el señor presidente. Buenas tardes, queridas y queridos. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω και να σας ευχηθώ καλό απόγευμα, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε, κύριε Επίτροπε, κύριε Υπουργέ. Μπορούμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με την απογευματινή μας ε, συνεδρίαση. Έχουμε τα όσα συνέβησαν χθε, τις ε, ψηφοφορίες, ε, τα κείμενα είναι έτοιμα αν κάποιος θέλει να τα σχολιάσει. Βλέπω πως δεν υπάρχουν όμως τέτοιες επιθυμίες, άρα λοιπόν μπορούμε τα πρακτικά της χθεσινής συνεδρίασης να τα εγκρίνουμε και να περάσουμε στο πρώτο σημείο της απογευματινής ημερήσιας συνεδρίασης που είναι οι δηλώσεις της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου για την πολιτική κατάσταση στη Ρουμανία. Θα ήθελα καταρχήν να σας ανακοινώσω πως με ιδιαίτερη ικανοποίηση έχουμε κοντά μας τον κύριο Στεφάνος Γκονέα που είναι πρόεδρος της Βουλής ε, της ε, Ρουμανίας και έχουμε και τον Υπουργό που είναι υπεύθυνο για τις σχέσεις με το Κοινοβούλιο στη χώρα αυτή. Θα ήθελα λοιπόν να τους καλωσορίσουμε ε, και τους δύο αυτούς επιφανείς επισκέπτες γιατί βέβαια θα παρακολουθήσουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την τόσο σημαντική συζήτηση που θα κάνουμε εδώ. Θα ήθελα να ξεκινήσω δίνοντας το λόγο στον κύριο Μαυρογιάννη, ο οποίος εξ του Συμβουλίου θα κάνει μια δήλωση για την κατάσταση στη Ρουμανία. Θα ήθελα να σας συγχαρώ και να συγχαρώ και την Προεδρία την Κυπριακή για την φιλοξενία που μας προσέφεραν